Invito a Προσκαλώ τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εκφωνήσει την ομιλία του, ο κύριος Αντώνιο Ταγιάννη. Μεγαλειότατη, κύριε Πρόεδρε, κύριοι Πρωθυπουργοί, συνάδελφοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων, κυρία Κόλ Ρίχτερ, μέλη της οικογένειας, εξοχότητες, και συμμετέχοντες και συμμετέχουσες σε αυτή την τελετή. Σήμερα αποτείουμε τον τελευταίο φόρο τιμής στο Χέλμουτ Κόλ. Έναν μεγάλο Ευρωπαίο, έναν μεγάλο κρατικό ηγέτη, έναν πολιτικό γίγαντα που ήταν ικανός να ακούει τους πολίτες και να βλέπει μακριά στο μέλλον. Ο Χέλμουτ Κόλ ήταν πάνω απ' όλα ένας άνθρωπος με κουράγιο, ένας θειασότης της ελευθερίας και της δημοκρατίας, πρωταγωνιστής στην επανένωση της Υπήρου μας. Προασπίστηκε την αξιοπρέπεια του ανθρώπου πάντοτε και σε κάθε μέρος του κόσμου, ενάντια στα τείχη, ενάντια σε κάθε είδους σιδηρούν παραπέτασμα, ενάντια σε κάθε πολιταρχισμό. Οι ιδρυτικές αξίες της Ένωσής μας υπήρξαν η σημαία και το λάβαρο των ε, πολυάριθμων αγώνων του. Οι ίδιες αξίες ενέπνευσαν και τη συνθήκη της Ένωσης. Ειρήνη, ελευθερία, ευημερία, ασφάλεια, δικαιοσύνη χωρίς σύνορα. Η βαθιά του πίστη σε αυτές τις αξίες, η βαθιά του πίστη στον άνθρωπο, ήταν η βάση της βαθιάς συμφιλίωσης μεταξύ ημών των Ευρωπαίων. Και αυτό άγγιξε τη μνήμη μας. Ο Χέλμουτ Κόλ ήταν ένας πρωταθλητής για μια γενιά που αφοσίωσε τη ζωή της στην καινούργια αναγέννηση στην Ευρώπη. Η τελευταία γενιά που έζησε στο πετσί της τον εφιάλτη του πολέμου. Για εκείνη τη γενιά η Ευρωπαϊκή Ενότητα, η υπέρβαση των εθνικισμών ήταν ακριβώς το όνειρο για ένα μέλλον ειρήνης για τα ίδια τους τα παιδιά. Σε αυτή τη γενιά ανήκε με όλη της την αξία και μια μεγάλη κυρία η Σιμών Βέιλ. Σήμερα θέλουμε να τιμήσουμε τη μνήμη της ε, σε αυτό το κοινοβούλιο και εκείνης Καθώ ήταν η πρώτη που προείδρευσε μετά τι εκλογέ με καθολική ψηφοφορία. Η ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον ήταν η πρώτη αρετή και δύναμη αυτών των μεγάλων Ευρωπαίων. Η ίδια ελπίδα που επέτρεψε πριν από αυτού στου ιδρυτέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Σούμαν, τον Τεγκάσπερη, τον Αντενάουερ, τον Σπακ, να επουλώσουν τι βαθιέ πληγέ που είχε αφήσει πίσω του ο πόλεμο. Χάρη σε εκείνου ξεφύγαμε από τι ηθικές και ε, υλικέ στάχτε που έχει αφήσει πίσω τη ε, η σύγκρουση. Μπορέσαμε να νοικοδομήσουμε και να επανενώσουμε την ήπειρό μα, φέρνοντα στο κέντρο των μεριμνών μα την ελευθερία και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Ο Χέλμουντ Κόλ αξίζει πέρα από κάθε αμφιβολία μια θέση τιμή στο πάνθεον των Ευρωπαίων. Το 1983, απευθυνόμενος στους Ευρωβουλευτές, είπε «Όποιος κοιτάξει την Ευρώπη μπορεί να αντιληφθεί πώς μπορεί το πεπρωμένο να βασίζεται στην φιλία και στη συνεργασία. Με αυτό το πνεύμα εργάστηκε άοκνα για να ενισχύσει την Ένωση, να την διευρύνει συμπεριλαμβάνοντας όλες τις δημοκρατίες της Επίρου και να ε, εδρεώσει την Ατλαντική Συμμαχία. Στα 16 χρόνια της θητείας του ως καγκελαρίου Κόλ ήταν πάντοτε πρωταγωνιστής καθοριστικός σε όλα τα γεγονότα. Δεν υπήρξε καμία σελίδα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που να μην έχει το αποτύπωμα της τόλμης του. Και σε αυτή την τόλμη οφείλουμε την ενίσχυση του ρόλου του Κοινοβουλίου, τη δημιουργία ενός μεγάλου χώρου ελευθεριών για τους πολίτες, πολιτικών και οικονομικών ελευθεριών, την γέννηση του κοινού την πολιτική της συνοχής. Γνώρισα τον καγκελάριο Κόλ όταν ως νέος πολιτικός το 1994 συνόδευσα τον Ιταλό Πρωθυπουργό σε επίσημη επίσκεψη στη Βόνη. Εντυπωσιάστηκα από το ταλέντο του, από την διορατικότητά του και την ε, διάβγεια από τον διέκρινε και τη δυνατότητά του να κατανοεί ακούγοντας τους άλλους και να σέβεται τι απόψει του. Για μένα ήταν σαφέ από τότε ότι για το Helmut Kohl η επανένωση σήμαινε πραγματικά όχι μια γερμανική Ευρώπη, μια Ευρώπη πιο γερμανική, αλλά μια Γερμανία που θα έπαιρνε πιο ευρωπαϊκό χαρακτήρα. Η επανένωση τη Γερμανία αλλά και τη Ευρώπη ήταν για εκείνον όπω και για τον Άντενάουερ δύο όψει του ίδιου νομίσματο. Η Ευρώπη του Κολ δεν δίστασε να τίνει τη χείρα στι νέε δημοκρατίε τη ε, Ανατολική Ευρώπη. Υπήρξαμε ένας φάρος ε, για την ελευθερία φέρνοντας κοντά μας εκατομμύρια Ευρωπαίων που έβγαιναν από τα σκοτάδια των κομμουνιστικών δικτατοριών. Για εκείνου η Ένωση άνοιξε τις ε, πύλες της με αλληλεγγύη, του συνόδευσε στην πορεία της ε, οικονομίας, της αγοράς, το κράτος δικαίου και την ευημερία. Η Ευρώπη του Κολ δεν είχε κανένα φόβο να σφυριλατήσει με νέε δυνάμεις το δικό της μέλλον. Ιδού, σε λίγα λόγια, το τεράστια, η τεράστια κληρονομιά που μας άφησε ο Κόλ, αλλά και η τεράστια ευθύνη που συνοδεύει αυτή την κληρονομιά. Αυτή η μεταλαμπάδευση ε, της κληρονομιάς του, όπως τις κυταλοδρομίες μιας κοιτάλη πρέπει να μας ε, δώσει το θάρρος να προχωρήσουμε. Στη διάρκεια της ζωής του, ο Χέλμουτ Κόλ έλαβε πολλές ε, τιμητικές διακρίσεις για τη συμβολή του στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση, μεταξύ αυτών το βραβείο Σαρλεμάνι, όπως και το βραβείο Πρίγκιπας των Αστουριών. Όμω η πραγματική αναγνώριση είναι αυτή που το επιφυλάσσει σήμερα η ίδια ιστορία. Περισσότερο από ποτέ το παράδειγμά του πρέπει να μας οδηγήσει για να συνεχίσουμε να οικοδομούμε από κοινού το μέλλον μας. Για να έρθουν πιο κοντά τα θεσμικά όργανα της Ευρώπης στους λαούς της Ευρώπης. Για να δώσουμε χειροπιαστές απαντήσεις στις ανησυχίες τους. Σήμερα περισσότερο από ποτέ πρέπει να διδαχτούμε από τον κόλ να διαλέξουμε την ελπίδα και να αφήσουμε κατά μέρο τον φόβο. Αυτό ακριβώς μας ζητούν και οι συμπολίτες μας. Το κουράγιο να είμαστε ενωμένοι, την τόλμη να αλλάξουμε, γιατί δεν είναι οι δυσκολίες ή τα προβλήματα που καθορίζουν τους Ευρωπαίους και τους ορίζουν την ταυτότητά τους, αλλά η δυνατότητά τους να τις ξεπερνούν. Όπως ο Κολ και οι άλλοι ηγέτες ε, του καιρού του πρέπει να εργαστούμε από κοινού για να αναθερμάνουμε το ευρωπαϊκό ιδεώδες. Μια Ευρώπη που είναι πιο αποτελεσματική, που μπορεί να προστατεύει τους πολίτες απέναντι σε αυτή την ε, θάλασσοταραχή που έχει γίνει η, η φίλιος. Όταν ε, διακυβεύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, ε, όταν υπάρχουν διακριτικές μεταχειρήσει κατά των ανθρώπων και βίες συμπεριφορέ κατά της πίστης τους, του δογματός τους τότε ο κόσμος στρέφεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ζητά ελπίδα και στήριξη. Αυτή η Ευρώπη, η δική μας Ευρώπη, πρέπει να σηκώσει το κεφάλι και να ξαναγίνει το σύμβολο των αξιών παντού στον κόσμο. Μια Ευρώπη που θα είναι πραγματικά φάρο που θα οδηγεί προ την ελευθερία. Μια Ευρώπη που θα προστατεύει τα δικαιώματα. Ο, ε, η μόνη ήπειρο όπου έχει καταργηθεί η θανατική ποινή. Ιδού τι Ευρώπη είχε επιθυμήσει ο Χέλμουντ Κόλ. Όχι απλώ μια αγορά ή ένα κοινωνόμισμα μια ταυτότητα που να έχει ε, πλαστεί μέσα από τους αιώνες, ε, το, την αίσθηση του ανήκειν σε μια κοινότητα, ένα ειδόδης ελευθερίας, ευημερία και ειρήνης. Στη Ρώμη στις 25 Μαρτίου του 2017, 60 χρόνια μετά την υπογραφή των συνθήκων, ε, δεσμευτήκαμε να συνεχίσουμε τη δουλειά του Κόλ και των άλλων μεγάλων Ευρωπαίων. Όπως έχουμε δείξει ως τώρα, θα πρέπει να κοιτάζουμε πέρα από τα κοντόφθαλμα συμφέροντά μας. Θα πρέπει να μας οδηγούν οι ηθικές αξίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η επανένωση της Γερμανίας είναι ένα από τα αναντήρητα παραδείγματα αυτής της πορείας. Το ίδιο και η υπέροχη χειρονομία φιλία και συμφιλίωση με τον Φρανσουά Μιτεράν στο Βερντά. Δύο άντρε, δύο λαοί, δύο έθνη που ε, συμφιλιώθηκαν στο ίδιο το μέρο όπου κάποτε είχαν έρθει αντιμέτωποι ω εχθροί. Δεν είναι ο πιο εύκολο δρόμο, ούτε ο πιο σύντομο. Όμω είναι ο μόνο δρόμο που μπορούμε να ακολουθήσουμε για να έχει μία έννοια ε, η ε, προσπάθεια αυτού του κοινού εγχειρήματο, του δικού μα εγχειρήματο, με ελπίδα και προοπτικέ για το μέλλον των επόμενων γενεών. Για όλους αυτούς τους λόγους η μνήμη του Κολ ήταν και θα παραμείνει ζωντανή στις καρδιές όσων, όπως όλοι εμείς, αγαπούν την Ευρώπη. Σε ευχαριστούμε, Χέλμουτ Κόλ. Ε, το δικό σου ιδεώδες για την Ευρώπη θα το ε, κουβαλάμε μαζί μας και στο μέλλον. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριο Ζόντο Κλοντ Γιούγκερ. Κύριε Πρόεδρε του Κοινοβουλίου, μεγαλειότατη, κυρίες και κύριοι Πρόεδροι, Κυρίε και κύριοι Πρωθυπουργοί, εξοχότατοι, κυρίε και κύριοι, αγαπητοί φίλοι που είστε πολλοί εδώ παρόντε, σήμερα που χαιρετούμε τον Χέλμοντ Κόλ, το Γερμανό και Ευρωπαίο ηγέτη. Εγώ αποχαιρετώ έναν πιστό φίλο, ο οποίος με συνόδευσε στοργικά επί έτη και δεκαετίες. Σήμερα δεν ομιλεί εδώ ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά ένας φίλος στο πρόσωπο του Χέλμουτ Κόλ μας ε, αφήνει ένας μεταπολεμικός γίγας. Ήδη εν ζωή είχε εγγραφεί στα ιστορικά εγχειρίδια, στα οποία θα παραμείνει για πάντα. Ήταν κάποιος που έγινε ένα μνημείο της Υπήρου, όπου καταθέτουν στεφάνι Γερμανοί και Ευρωπαίοι, οφείλουν να καταθέτουν. Ήταν δική του επιθυμία να τον αποχαιρετήσουμε εδώ στο Στρασβούργο σε τούτη εδώ τη γαλλογερμανική πόλη. Μια ευρωπαϊκή μεθόριο. Πόλη την οποία αγάπησε και έπρεπε να τιμηθεί ε, η ιδέα του. Δεν είναι γερμανική σημερινή τελετή, αλλά είναι ευρωπαϊκή και γερμανική. Αρχίζει η μέρα σήμερα στο Στρασβούργο και τελειώνει στο Σπάιε. Ε, στο καθεδρικό ναό, σε μια πόλη που αγαπούσε. Ο Χέλμουντ Κόλ ήταν Γερμανός πατριώτης, αλλά και Ευρωπαίος πατριώτης. Ήταν κάποιος που έφερνε κοντά και ένωνε τους ανθρώπους και τα πράγματα. Ένας Γερμανός και Ευρωπαίος πατριώτης μάλιστα, διότι για εκείνον δεν υπήρχε αντίφαση ανάμεσα στο τι είναι γερμανικό και τι είναι ευρωπαϊκό, τι οφείλει να είναι ευρωπαϊκό. Ο Γάλλος φιλόσοφος Πασκάλ είχε πει ότι του αρέσουν τα πράγματα που ταιριάζουν μεταξύ τους, που συμβαδίζουν. J'aime les choses Για το Helmut Kohl συμβάδιζαν η γερμανική και η ευρωπαϊκή ενοποίηση. Δύο όψεις του ιδίου νομίσματος, όπως άλλωστε και ο Adenauer και ο ίδιος. Αυτό το αξίωμα του Adenauer το υιοθέτησε και με τη δράση του και τη σκέψη του το μετέφερε στην πράξη. Συνέχεια. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα γι' αυτό. Η πτώση του τείχους του Βερολίνου. Έγινε δεκτή παγκοσμίω αλλά και στην Ευρώπη με χαρά. Η Γερμανική Επανένωση, την οποία ανυποχώρητα πίστευε, γνώρισε όμως ε, αντιδράσεις και αντιστάσεις και ανοιχτή απόρριψη πολλές φορές στην Ευρώπη. Σε πολλές συνομιλίες υπομονετικές ε, και κατηδίαν φρόντισε να προωθήσει τη Γερμανική Επανένωση. Και είχε επιτυχία σε αυτό γιατί η φήμη του, την οποία είχε κατακτήσει από χρόνια, του επέτρεπε να το κάνει και να αποδείξει ότι φιλοδοξούσε να είναι Ευρωπαϊκή Γερμανία και όχι Γερμανική Ευρώπη. Με όλες του τις δυνάμεις θέλησε την επανένωση της Γερμανίας και έπεισε και άλλους εκτός Γερμανίας, κατάφερε να το κάνει, ότι ήταν ιστορικά σωστός αυτός ο δρόμος κατάφερε να καταλάβει ότι έπρεπε να δράξει το μανδύα του Θεού που κοιμάτιζε για μια σύντομη στιγμή πάνω από την ιστορία. Αυτό δεν το αντελήφθηκαν αμέσω όλοι στην Ευρώπη. Την κίνηση αυτή του μανδύα του Θεού. Εκείνο ναι. Ένιωσε ότι ήταν κοντά, ότι μπορούσε να αγγίξει τη γερμανική ενοποίηση. Κατάφερε να γνωρίσει και να αξιοποιήσει την εύνοια των καιρών. Άλλοι θα είχαν αποτύχει σε αυτή την ιστορική στιγμή και πραγματικά καταλάβαμε ότι ήταν διορατικός. Ο Χέλμουντ Κόλ σκεφτόταν τη Γερμανία, αλλά ε, η προοπτική του ήταν στην Ευρώπη και πάντα το βλέμμα του στραμμένο προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Όχι μόνο προς την Πολωνία, αλλά ιδιαίτερα προς την Πολωνία. Ο, Κόλ δεν ήταν υπεύθυνο για τα εγκλήματα των Ναζί στην Πολωνία, αλλά είχε επίγνωση της ιστορικής ευθύνης που ευάρυνε τη Γερμανία. Όπως και ο Βίλι Μπραντ, ε, με τον οποίο ε, συνδέθηκε πολύ στο τέλος της ζωής του. Δύο σπουδαίοι άνδρες της εποχής μας, ο Κολ και ο Μπραντ. Η διεύρυνση προς Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη χωρίς την Πολωνία ήταν κάτι το οποίο ε, ήταν απλώς τα αδιανόητο για τον Κολ και θα ήταν πραγματικά πολύ επιθυμητό να μην ξεχνάμε κάτι τέτοιο. Ο Χέλμουτ Κόλ δεν ήταν μόνο αρχιτέκτονας γερμανικής ενοποίησης. Πολύ περισσότερο από άλλοι βοήθησε σημαντικά για τη συμφιλίωση ανάμεσα στην ευρωπαϊκή ιστορία και την ευρωπαϊκή γεωγραφία. Είναι μεταξύ εκείνων που κατάφερε να τερματίσει τη διχαστική συμφωνία της Γιάλτας για την Ανατολική και Δυτική Ευρώπη. Και η Νότια Ευρώπη, όχι μόνο Ανατολική και Κεντρική, οφείλουν πολλά τον κόλ και θα πρέπει να το θυμόμαστε αυτό. Επίσης, προώθησε τις σχέσεις με το Ισραήλ και τις μεταξέλιξε και με την καρδιά και με τον νου. Ήταν μέγας φίλος του Ισραήλ. Επίσης, βοήθησε να βελτιωθούν οι σχέσεις ε, με την πρώην Σοβιετική Ένωση και την ε, Ρωσική Ομοσπονδία. Ο ιστορικός Κόλ και ο καγκελάριος Κόλ γνώριζε το ποικίλο βάθος της Ρωσίας και ταυτόχρονα ήταν πεπισμένος ατλαντιστής και ε, δραστήριος μάλιστα. Μετά το Χέλμουντ Σμιτ επέβαλε τη διπλή απόφαση του ΝΑΤΟ κόντρα στα τότε σημεία των καιρών. Μάικε, φίλοι, ίσως είμαι ο μόνος εδώ στην αίθουσα που έχω δει τον Χέρμουτ Κόρ να κλαίει σε συνεδρίαση στις 13 Δεκεμβρίου 1997. Εκείνη τη μέρα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπό την Προεδρία μου στο Λουξεμβούργο αποφάσισε τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη αλλά και την Κύπρο και τη Μάλτα. Κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματο, ζήτησε το λόγο κατ' εξαίρεση το ζήτησε, γιατί συνήθω μιλούσε χωρί να ζητήσει το λόγο. Ζήτησε το λόγο λοιπόν κατά τη διάρκεια του γεύματο και είπε με φωνή πνιγμένη από τα δάκρυα ότι αυτή η μέρα τη έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων ε, ήταν από τις πιο ωραίες στιγμές της ζωής του. Εκείνο ω Γερμανός καγκελάριο ότι είχε την ευκαιρία αυτή τη ιστορική στιγμή να ζήσει την Ευρώπη να πορεύεται μαζί. Αυτό τον γέμιζε με μεγάλη συγκίνηση την κάθε εκμάδα του. Μετά από όλα αυτά τα δεινά στα οποία έχει επιβάλει την Ευρώπη η Γερμανία. Μετά σταμάτησε. Συλλογισμένος κάθισε και έκλαιγε πολλά λεπτά και δεν ήταν ο μόνος. Και κανείς τότε δεν τράπηκε που έκλαιγε. Καλύτερες στιγμές της Ευρώπης. Europe at its best. Ακόμα και για το ευρώ, μαζί με το φίλο μου τον Τέο Βάιγκελ, ήταν η κινητήρια και η φέρουσα δύναμη. Σίγουρα, αμήλικτα, ε, ήξερε να εκπροσωπεί τα γερμανικά συμφέροντα. για την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Στην αρχή το ζήτησε φιλικά και μετά το επέβαλε ε, ε, με επίταση. Και χωρίς τον κόλ δεν θα υπήρχε σήμερα το ευρώ η νομισματική ένωση στα μάτια του έκανε μία αναστρέψιμη την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Για εκείνον το ευρώ παρέμενε ευρωπαϊκή νευτική πολιτική με άλλα μέσα. Και κάτι άλλο που χαρακτηρίζει τον κόλ. Σεβόταν με τον ίδιο τρόπο όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεγάλα και κυρίως τα μικρά κράτη-μέλη. Αισθάνονταν ότι τα καταλάβαινε και ότι συμμεριζόταν τα συμφέροντά τους. Και ένα τελευταίο. Στην Ευρώπη συμβαίνει συχνά. Όταν κινδύνευαν να αναβαγίσουν οι διαπραγματεύσεις, τότε έβγαινε ο κόλ εμπρός και μας επέπλητε στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για να μην αναλωνόμαστε σε εθνικούς εγωισμούς. Κύριε Πρόεδρε της Γαλλικής Δημοκρατίας, τέλος, ο Χέλμουτ Κόλ ήταν ο άνθρωπος της συνέχισης της γαλλογερμανικής συμφιλίωσης. Με σθένος και θέρμη συνέχισε το έργο των Ντεγκόλ και Άντεναουαρ. Εκείνος που δεν μιλούσε γαλλικά, ήξερε τα πάντα για τη Γαλλία, για την ιστορία της, για την ε, βαθιά Γαλλία, τις περιφέρειες, ιδιαίτερα για την Αλσατία, την οποία αγαπούσε, ε, επισκεπτόταν συχνά τη λάτρευε και ήξερε και τα καλά εστιατόρια της Αλσατίας που είναι και πολλά. Η, ιστορία θα κρατήσει μια εικόνα που λέει τα πάντα για τον Κόλ και τη στενή σχέση που είχε με τη Γαλλία. Την ημέρα που στο Βερντά ο Χέλμοντ Κόλ και ο Φρανσουά Μιτεράν έδωσαν το χέρι ένα στον άλλο. Εσφράγισαν εκείνη τη μέρα για πάντα την αδελφοσύνη ανάμεσα στη Γαλλία και τη Γερμανία. Το γεγονό ότι τον αποχαιρετούμε σήμερα εδώ στο Στρασβούργο, στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που ήταν πάγιος φίλος, δίπλα στο Ρήνο, που είναι τόσο γεμάτος ιστορία και τραγωδία για την Ευρώπη και σύμβολο. Σε αυτή την ωραία πόλη του Στρασβούργου, για την πρωτεύουσα, μία από τις πρωτεύουσες της Ευρώπης, είναι σημαντικό να τιμά σήμερα τη μνήμη του Ευρωπαίου Χέλμουτ Κόλ. Μάλιστα, ο Χέλμουτ Κόλ ήταν Γερμανός και Ευρωπαίος πατριώτης. Ο πατριωτισμός για εκείνον δεν ήταν ποτέ ένας πατριωτισμός απέναντι σε κάποιους άλλους, αλλά ένας πατριωτισμός που, που με κάποιους άλλους. Η Ρινανία Παλατινάτο, η Γερμανία και η Ευρώπη υποκλίνονται σήμερα ε, μπροστά στην εντυπωσιακή ζωή και το έργο του Χέλμουτ με ευγνωμοσύνη και με δέος. Ήταν γεμάτη η ζωή του. Θα έχει ξεχάσει ορισμένε αντικσότητες, αλλά πολλά θα θυμάται ακόμα. Γνωρίζει και εμείς το ξέρουμε και ε, άλλωστε ότι έχει βελτιώσει την Ευρώπη. Αγαπητέ Χέλμουντ, ελπίζω, πιστεύω να είσαι στον παράδεισο. Θα προτιμούσαμε να είσαι εδώ. Ε, να μου υποσχεθείς ότι δεν θα σπεύσεις στον παράδεισο να ιδρύσεις ε, τοπική οργάνωση της Τσέντεου. Έχεις κάνει αρκετά για το κόμμα σου, για τη χώρα σου και για την κοινή μας Ευρώπη. Σε ευχαριστώ πολύ, Χέλμουτ. Αναπαύσω εν ειρήνη, καγκελάριε και αγαπητέ φίλε. Μετά από τη γεμάτη και πλούσια ζωή σου, κέρδισες αυτή την ειρήνη. Αιωνία σου η μνήμη. Merci, Σας ευχαριστώ. Καλώ τον κύριο Ντόναλτ Τούσκ, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, να εκφωνήσει την ομιλία του. Μεγαλειότατη. Αγαπητά μέλη της οικογένειας, κυρίες και κύριοι, ως Ευρωπαίος, ως Πόλωνος και ως κάποιος που κατάγεται από το Κτάνσκ εξίσου, θεωρώ πως βρίσκομαι σε πολύ καλή θέση για να πω λίγα λόγια για να αποχαιρετήσω τον Χέλμουτ Κόλ, επίτιμο πολίτη της Ευρώπης και επίτιμο πολίτη του Γκτάνσκ. Δεν είναι τυχαίο το ότι η γενέτειρά μου, η πόλη στην οποία γεννήθηκε το Συνδικάτο της Αλληλεγγύης, αποφάσισε να κάνει τον καγκελάριο Κόλ επίτιμο πολίτη της. Λίγοι άνθρωποι στην Ευρώπη αντιλαμβανόταν πόσο σημαντική ήταν για την ελευθερία η εξέγερση σε διάφορες πόλεις στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη για την ιδέα της Ενωμένης Ευρώπης. Πολλές φορές μας υπενθύμιζε πως οι πρώτοι οι οποίοι ράγισαν το τείχος του Βερολίνου ήταν οι άνθρωποι που δούλευαν στα ναυπηγεία του Γκτάνσκ το 1980. Και γι' αυτό ακριβώς ο καγκελάριος Κολ προώθησε την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση των χωρών που ανήκαν στο Σοβιετικό μπλοκ. Έχει μεγάλη ιστορική σημασία και συμβολική το ότι ο Χέλμουτ Κόλ έμαθε την πτώση του τείχους του Βερολίνου. Όταν ήταν σε επίσκεψη επίσημη στην Βαρσοβία, είχε επισκεφθεί τον πρώτο μη κομμουνιστή πρωθυπουργό. Και εκεί πέρα, στην Βαρσοβία, μίλησε για πρώτη φορά για την ιδέα της Ενωμένης Γερμανίας. Από την Βαρσοβία, την πόλη που είχε υποφέρει τόσα πολλά από τους Γερμανούς στον Δεύτερο Παγκόσμιο. Στην διαδικασία αυτή της συμφιλίωσης, ο Χέλμουτ Κόλ συνεισέφερε πάρα πολύ. Χάρη σε αυτόν, μεταξύ άλλους, απέκτησαν νόημα ξανά λέξεις όπως η εμπιστοσύνη και η συμφιλίωση, ειδικά στις γαλλογερμανικές και τις γερμανοπολωνικές σχέσεις. Θυμάμαι ακόμα δύο πολύ ισχυρές εικόνες. Τον πρόεδρο Μιτεράν και τον καγκελάριο Κολ χέρι-χέρι στο Βερντέν και τον Πρωθυπουργό Μαζοβιέτσκι και τον καγκελάριο Κολ αγκαλιασμένους στην Κεζόβα δύο μέρες μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου. Οι χειρονομίες αυτές και οι αποφάσεις που ακολούθησαν έθεσαν τα θεμέλια της σημερινής Ευρώπης. Ο Χέλμουτ Κόλ μετέφρασε σε πολιτική πράξη τα λόγια του Τόμας Μαν. ότι θέλουμε μια ευρωπαϊκή Γερμανία, όχι μια γερμανική Ευρώπη. Όμως, το όραμά του και η ματιά του απλωνόταν πέρα από τα σύνορα της Γερμανίας. Με εξαιρετική αποφασιστικότητα προσπάθησε να ορίσει μια κοινή Ευρώπη. Αναζήτησε τα όσα μας ενώνουν και όχι τα όσα μας χωρίζουν, χωρίς να τρέχει ψευδεστήσεις ότι θα ξεπεραστούν έτσι εύκολα. Υπάρχει σήμερα μια ενωμένη Ευρώπη γιατί βρήκε εταίρους σε αυτή τη μεγάλη προσπάθειά του. Τους γίγαντες της ευρωπαϊκής πολιτικής, τον Λέχ Βαλέσα, τον Φρανσουά Μιτεράν, τον Ταντέους Μαζοβιεύσκη, τον Βάτσλαβ Χάβελ και σε μια διαφορετική διάσταση τον Πάπα Ιωάννη Παύλο τον Δεύτερο. Σήμερα οι διάδοχοι των μεγάλων αυτών ηρώων της θετικής ιστορίας της Ευρώπης πρέπει, καθώς βρίσκονται εδώ συγκεντρωμένοι γύρω από αυτό το φέρετρο, να εξετάσουν τη συνείδησή τους. Στο Βερολίνο, στη Βαρσοβία, στο Παρίσι και στη Βουδαπέστη, το ερώτημα για το μέλλον της Ενωμένης Ευρώπης πρέπει να απαντηθεί με ένα δυνατό ναι. Ναι στην Ένωση, ναι στην ελευθερία, ναι στα ανθρώπινα δικαιώματα. Στο τέλος της θείας λειτουργίας της συμφιλίωσης στην Κριζόβα, ο καγκελάριος Κόλλη είχε πει τότε. Ας πάμε προς το ιερό αυτό, προς ένα ειρηνικό μέλλον, ευλογημένο από τον Θεό, για τους λαούς μας, για τους λαούς της Γερμανίας και της Ευρώπης, για όλους μας στην Ευρώπη. Αυτά τα λόγια θα ήθελα να μείνουν στη μνήμη μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τώρα θα δούμε την ταινία «Χέλμουτ Κόλ, ένας σπουδαίος Ευρωπαίος. Μόνο μια ενωμένη, ισχυρή και ενωμένη μπορεί σε συνεργασία με τους φίλους και συμμάχους στη Βόρεια Αμερική και σε απαραίτητο διάλογο με την Ανατολή να βρει ε, μια ισορροπία που είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη της ειρήνης παγκοσμίως. Στην ε, Ανατολική Γερμανία, στο Βερολίνο, έχουμε ξεπεράσει ειρηνικά το τείχος και τα καθοτά πλέγματα. Μετά από 30, 30 ε, έτη ε, του διχασμού, ο κόσμος εορτάζει την ενότητα, το συνέστημα του ανήκειν, Χρειαζόμαστε μια ισχυρή Ευρώπη και Ευρώπη με αυτοπεποίθηση. Αν δεν θέλουμε να γίνουμε το μπαλάκι της παγκόσμιας πολιτικής. Το επαναλαμβάνω, όλοι χρειαζόμαστε την Ευρώπη. Στο 19ο αιώνα ήταν τα εθνικά κράτη. Αυτά δεν μπορούν να διαβούν το κατόφλι του 21ου αιώνα. Στις νέες δημοκρατίες στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη γίνονται μεταρρυθμίσεις προς το καλά νοούμενο συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παντού όπου κανείς διαβαίνει απρόσκοπτα τα σύνορα, που ανταλλάσσει ιδέες και απόψεις ελεύθερα, όπου οι άνθρωποι μπορούν να συναντούν το ένα στον άλλον, η έχθρα και η καχυποψία δεν ευδοκιμούν. Και η καλύτερη εγγύηση μια, για μια βιώσιμη και ασφαλή ειρήνη στην Ευρώπη είναι και παραμένει η ελευθερία των ανθρώπων. Παρακαλώ τον κύριο Φελίπε Γκονθάλεθ Μάρκεθ, πρώην Πρωθυπουργό του Βασιλείου της Ισπανίας, να έχει την καλοσύνη να πει δύο αποχαιρετιστήρια λόγια. Ευχαριστώ τους Προέδρους του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου που μου κάνουν αυτή τη τιμή. Ευχαριστώ και την σύζυγο του κ. Κόρ. Μου δίνει την ευκαιρία να χαιρετήσω ένα φίλο μου προσωπικά και να τον αποχαιρετήσω. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε μόνο πέντε λεπτά γιατί μου στοιχίζει πολύ. Αποχαιρετώ το Helmut Κόλ. γιατί είχαμε φιλία βαθιά με εμπιστοσύνη. Είναι σπάνιο είδος αυτό στις πολιτικές σχέσεις και ήταν και πιστός και φίλος και όταν έλειπε αυτή η πίστη και αφοσίωση ήταν πολύ ευαίσθητος αυτό. Είχε συνείδηση της ιστορίας, γι' αυτό μιλούσε για ευρωπαϊκή Γερμανία, για να μην ξαναζήσουμε ποτέ μια γερμανική Ευρώπη και είχε και αίσθημα για τα κοινωνικά. Κάποιοι το ξεχνούν αυτό. Επίστευε στην κοινωνική οικονομία της αγοράς. Και ποτέ δεν θεώρησε ότι η κοινωνική διάσταση της ευρωπαϊκής οικοδόμησης ήταν μια πρόφαση ή ένα εμπόδιο για την ένταξη της Ευρώπης στην πακοσμιοποίηση. Μεγαλειότατη, εξοχότατη αρχηγή κρατών και κυβερνήσεων. Χάνουμε ένα μεγάλο ευρωπαϊστή και έχω την αίσθηση ότι έχασα ένα φίλο με τον οποίο συμμεριζόμουν και συμμερίστηκα ιστορικές, αποφασιστικές στιγμές για τη Γερμανία, για την Ισπανία, για την Ευρώπη και για τον κόσμο ολόκληρο. Από εκείνη την απόφαση στην οποία αναφέρθηκε προηγουμένως ο κύριος Γιούνκερ για τους πυράβλους μέσου βεληνικούς, όπου έδωσε μεγάλη μάχη, στην οποία ήμουν στο πλευρό του μέχρι που αρνήθηκε την ανάπτυξη και τον εξυγχρονισμό ε, των πυράβλων βραχαίους βεληνικούς. Και φυσικά μιλούσε γαλλικά. Μία φράση ήξερε στα γαλλικά. Όταν έπαιρνε το λόγο Φρανσό Μιτεράν, έλεγε «Il parle François Premier Legrand». Ομιλεί ο Φραγκίστος ο πρώτος, ο Μέγας, που ήταν ένας βασιλιάς της Γαλλίας. Μετά τις αποφάσεις όμως αυτές, μας βοήθησε πάρα πολύ με αλληλεγγύη για να ενταχθεί η Ισπανία στις ευρωπαϊκές τότε κοινότητες. Από κοινού, μαζί με τον Μιτεράν και τον Τελόρ και με άλλους φίλους, εορτάσαμε την υπογραφή της ενιαίας πράξης, που ήταν άμεσος προάγγελος ε, του μεγάλου βήματος της υπογραφής της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και μεσούσης αυτής της περιπέτειας και των μεγάλων ιστορικών προκλήσεων έπεσε το τείχος του Βερολίνου και κατάφερε να καλπάσει επάνω στο άλογο που έριξε το τείχος για να ενώσει τη Γερμανία η οποία αυτή η επανένωση είναι ενταγμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήθελε μια Ευρωπαϊκή Γερμανία, επαναλαμβάνω, ποτέ πια μια Γερμανική Ευρώπη. Αυτό τον καθορίζει και καθορίζει και τη βούλησή του. Και πίσω από αυτή την αντίληψη δέχτηκε το ευρώ με κίνδυνο να χάσει το αξίωμά του. Το ευρώ δεν ήταν μια νομισματική πράξη. Ωραία, είχαμε υπογράψει για την ΟΝΕ, αλλά γνώριζε ότι η εγκατάλειψη του Μάρκου μπορεί να του στήχιζε το αξίωμά του και το διακινδύνευσε. Εκείνη τη στιγμή όπου κάποια στιγμή έχασε τις εκλογές, κάποια στιγμή τις χάνουμε τις εκλογές όλοι μας. Λοιπόν, όταν έχασε τις εκλογές, του έλεγα, Χέλμουτ, με εκατομμύρια ψήφους κυβερνάς, αλλά για να ζήσεις χρειάζεσαι την αγάπη, τη στοργή, την εκτίμηση πολύ λίγων φίλων. Ακόμα είναι πιο σημαντικό να ζεις παρά να κυβερνάς. Όσο σημαντικό και να είναι να κυβερνάς. Εσύ έχεις καλούς και πιστούς φίλους για να σε συνοδεύουν στη ζωή. Σήμερα ένας από τους φίλους αυτούς, πιστός φίλος, θέλει να σας αποχαιρετιστεί και να πω ότι θα αφήσει πολιτικό κενό, μέγα πολιτικό κενό, το οποίο θα γεμίσει η θύμησή σου, η αποφασιστικότητά σου και μια πραγματική ιστορική αναφορά για τη ζωή και το έργο σου αλλά κυρίως για ανθρώπους όπως εγώ, θα αφήσει ένα μεγάλο κενό μιας μακράς φιλίας που δοκιμάστηκε σε σημαντικές ιστορικές στιγμές και μας αφήνεις μια στιγμή που σε χρειαζόμαστε. Δεν πρόκειται να σε ξεχάσουμε, Χέλμουτ. Μπορείς να υπολογίζεις τη φιλία μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Προσκαλώ τον κύριο Μπιλ Κλίντον, πρώην πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, να πει λίγα αποχαιρετιστήρια λόγια. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να πω λίγα λόγια. Ευχαριστώ τον Πίτερ, τον Βάλτερ, την οικογένεια του Χέλμουτ. Αγαπητοί ηγέτες Ευρώπης, ε, καγκελάρια, ε, κυρία Μέρκελ, ε, κύριε Μακρόν, Σας... Ε, θα ήθελα να σας πω να σκεφτείτε κάτι. Δεν είναι, διαβάζω εκτός... Μιλάω εκτός σημείωσεων. Θέλω να σας πω το εξής. Κοιτάξτε γύρω σας. Όλοι εμείς είχαμε αξιώματα. Και ήρθαμε εδώ. Ήρθαμε γιατί. Γιατί ο Χέλμουντ Κόλ μας έδωσε την ευκαιρία να εμπλακούμε σε κάτι μεγαλύτερο από τους εαυτούς μας, μεγαλύτερο από τις θητείες μας, μεγαλύτερο από τις σταδιοδρομίες μας. Γιατί όλοι αργά ή γρήγορα σε ένα τέτοιο φέρετρο θα καταλήξουμε. Και το μόνο δώρο το οποίο μπορούμε να αφήσουμε πίσω είναι ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας και την ελευθερία να κάνουν τις δικές τους επιλογές και τα δικά τους λάθη. Τον αγαπούσα. Η Χίλαρη λέει ότι τον αγαπούσα γιατί ήταν ο μόνος άνθρωπος που έτρωγε περισσότερο από μένα. ερχόταν τόσο συχνά στην Ουάσιγκτον που μία φορά με πήγε στο δικό του αγαπημένο εστιατόριο στην ε, Ουάσιγκτον. Ε, Φίλεμιν λέγεται, είναι ακόμα, μπορείτε να πάτε, είναι πολύ καλό. Γιατί τα λέω αυτά. Γιατί ο 21ος αιώνας στην Ευρώπη, όπως λέτε, ξεκίνησε στην δικιά του θητεία. Γιατί είχε να απαντήσει κάποια μεγάλα ερωτήματα τα οποία όλα έχουν επιπτώσεις σήμερα. Και επειδή λόγω των απαντήσεων που έδωσε σε αυτά τα ερωτήματα βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Θα πρέπει να υπάρξει πραγματικά ενωμένη Γερμανία μετά την πτώση του τείχους. Τι σημαίνει αυτό, πόσο θα κοστίσει, θα είναι δύσκολο. Αλλά είμαστε ένας λαός και μία χώρα και θα πρέπει να υποστούμε τις δυσκολίες και τις ταλαιπωρίες. Ακόμα και στην δική του την περίπτωση, ε, ακόμα και αν του κόστισε τις εκλογές. Γιατί χρειάστηκε βεβαίως πολύ περισσότερος χρόνος να εξισωθεί το ανατολικό κομμάτι από όσο είχε προβλέψει. Το άλλο ερώτημα είναι, εάν θα πρέπει να υπάρξει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να επεκταθεί ώστε η Γερμανία να μην είναι ξανά στο άκρο της Ευρώπης. Οι Πολωνοί, οι Ούγγροι, οι Τσέχοι και λοιποί. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό από κοινού. Θα πρέπει η Γερμανία που την αντιμετώπισαν οι γείτονές της με δυσπιστία να κινητοποιηθεί στρατιωτικά για να σταματήσει την σφαγή στην Βοσνία και να υποστηρίξει την πρώτη επέμβαση του ΝΑΤΟ εκτός των κρατών μελών του και την πρώτη ανάπτυξη γερμανικού στρατού στο εξωτερικό από τον Δεύτερο Παγκόσμιο και μετά. Μετά από όλες τις σφαγές του πολέμου τελικά όταν έπεσε το τείχος του Βερολίνου θα πρέπει να ανακουφιστούμε ή να αναγνωρίσουμε ότι πρόκειται για μια τρομερή εμπειρία για τη Ρωσία και να απλώσουμε ένα χέρι φιλίας και με μια επιταγή βεβαίως στο χέρι αυτό και να μου δώσει και εμένα την ευκαιρία να κάνω το ίδιο. Θα πρέπει να διατηρηθεί ή να καταργηθεί το ΝΑΤΟ. Πολλοί έλεγαν τότε ότι έπρεπε να καταργηθεί και ανταυτού επεκτάθηκε, όχι ως μια απειλή, αλλά ως υπόσχεση με μια σειρά εταιρικών σχέσεων που περιλαμβάνουν και την Ρωσία και την Ουκρανία για να εγγυηθεί την εδαφική ακαιρεότητα και την συνεργασία των χωρών στο μέλλον. Αυτά ήταν πραγματικά μεγάλα ερωτήματα. Τώρα ακούγεται εύκολο και λέμε όχι μόνο ήταν εύκολο, αλλά και κοιτάξτε πώς έχει διαμορφωθεί σήμερα η πραγματικότητα. Μπορεί όλοι εμείς τώρα να φαινόμαστε μικροί μπροστά στις τωρινές πραγματικότητες, αλλά δεν υπάρχουν μόνιμες νίκες ή ήττες στην πολιτική. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι το κίνητρό μας. Εγώ τον αγαπούσα αυτόν τον άνθρωπο γιατί η όρεξή του δεν σταματούσε το φαγητό. Γιατί ήθελε να δημιουργήσει έναν κόσμο στον οποίο κανείς δεν θα κυριαρχούσε. Έναν κόσμο στον οποίο η συνεργασία ήταν προτιμότερη από τη σύγκρουση και στον οποίο διάφορες ομάδες κάνουν, λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις από μεμονωμένους δικτάτορες ένα κόσμο στον οποίο οι νέοι μπορούν να πούν ότι εμείς κάναμε λάθος. Τέλο πάντων, αυτό το οποίο κάναμε εμείς μπορεί να μην αρκεί για τώρα. Όλα αυτά φανήκαν ακριβώς στο πώς αντιλαμβανόταν το μεγάλο βάρος που είχε η Γερμανία όταν ακριβώς έλαβε την απόφαση να μην έχει πλέον τον έλεγχο του νομίσματός της και τη δική της κεντρική τράπεζα. Ήταν κάτι το φυσικό. Σήμερα λοιπόν είμαστε σε μια εποχή πολιτικής που βασίζεται στην ταυτότητα. Το ποιοι είμαστε. Θα πρέπει να μας καθορίζουν περισσότερο οι διαφορές μας ή τα κοινά μας σημεία. Μην έχετε καμία αμφιβολία. Ο Χέλμουντ Κόλ πραγματικά ήταν πάρα πολύ ικανοποιημένος που ήταν α, ε, Γερμανός. Και όταν είχε έρθει στις Ηνωμένε Πολιτείες τον πήγα στο Μιλγουόκι σε ένα σχολείο γερμανικών και μίλησε εκεί πέρα με Αφροαμερικανούς μαθητές που έκαναν σχολείο στα γερμανικά. Αυτός έλεγε πως σε έναν εξαρτούμενο κόσμο, όπου τα, δίχτυα, τα σύνορα μοιάζουν περισσότερο με δίχτυα παρά με τείχους, όπου η τεχνολογία μας έκανε πιο συνδεδεμένους, αλλά και πιο ευπαθείς ε, στην τρομοκρατία, στην κυβερνοτρομοκρατία, ότι έπρεπε να αναζητήσουμε κοινά στοιχεία. Του άρεσε που ήταν Γερμανός. Μου έδινε να φάω κάτι πράγματα, δεν μου άρεσαν και πολύ γιατί ήταν Γερμανός και του άρεσε. Ήταν και Ευρωπαίος και του άρεσε. Αλλά με στην διάρκεια αυτής της μεγάλης ηγετικής του πόριας είχε αντιληφθεί ότι η καρκίνη του 20ου αιώνα γεννήθηκαν από ανθρώπου που θεωρούσαν ότι η κυριαρχία είναι καλύτερη από τη συνεργασία. Γι' αυτό βρισκόμαστε όλοι εδώ σήμερα. Όλοι μας γέροι άνθρωποι που ήρθαμε να το πούμε σας ευχαριστούμε που μας έδωσε την ευκαιρία να γίνουμε κάτι μεγαλύτερο από τους αυτούς μας. Να συνεισφέρουμε, να θυμόμαστε το τι έκαναν οι Πολωνοί εργαζόμενοι στο Γκτάνσκ. Η πολιτική τελικά αναφορά μεγάλες περιόδους κυριαρχίας, αλλά την δυνατότητα να ζήσουν καλύτερη ζωή όσο δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι. Και οι πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο μέρα σε ένα φέρετρο θα βρεθούν. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος είτε σκοτώσει είτε προστατεύει ζωές τελικά εκεί θα βρεθούν εκεί θα επιστρέψουν οι Αφροαμερικανείς εκκλησίες τους, τις κηδείες τις λένε επιστροφή εκεί θα γυρίσουμε όλοι Αλινόστηση. καλώς σου κατεβόδιο λοιπόν φίλε μου και το μεγαλύτερο δώρο που μας έκανες ήταν τα μαθήματα που έδωσες, ότι αυτό το οποίο έχει σημασία είναι το τι αφήνουμε στα παιδιά μας. Ελευθερία, ειρήνη, ασφάλεια. Για να μπορέσουν να επιδιώξουν τα δικά τους όνειρα. Και η πεποίθηση ότι μπορούμε να είμαστε μεγάλοι εξυψώνοντας. Καλά τα πήγες στη ζωή σου και υποκλεινόμαστε μπροστά σου. Thank you, Mr. President. Ευχαριστούμε, ο πρόεδρος, ε, πρόεδρος της ε, κυβέρνησης της ε, Ομοσπονδίας της Ρωσίας, να πάρει το λόγο. Уважаемая госпожа Коль Рихтер, κυρία Κόλ Ρίχτερ, συγγενής του Χέλμουντ Κόλ, κυρίες και κύριοι, σήμερα αποχαιρετούμε τον Χέλμουντ Κόλ, τον άνθρωπο που δικαίως αποκαλείται όχι μόνο ο αρχιτέκτονας της επανένωσης της Ευρώπης, αλλά και ο αρχιτέκτονας της Ενωμένης Ευρώπης και για να είμαστε και πιο άμεση ο αρχιτέκτονας του σημερινού κόσμου. Ο Χέλμουτ Κόλ ήταν μεγάλη προσωπικότητα με κάθε έννοια της λέξης. Ένας άνθρωπος με μεγάλα σχέδια, μεγάλες ιδέες. Ήταν ένας ηγέτης χάρη στον οποίον άλλαξε η εποχή του. Πολλά από τα πράγματα τα οποία πέτυχε στην 16η θητεία του ως καγκελάριος έλεγαν οι σύγχρονοί του ότι είναι αδύνατον να γίνουν. Σήμερα βεβαίως τα βλέπουμε διαφορετικά. Φαίνεται ότι δεν ήταν δυνατόν να γίνει κάτι διαφορετικό. Κατά το οποίο σημαίνει ότι επέλεξε την μόνη σωστή πορεία και διαμόρφωσε την ιστορία. Από αυτήν την έννοια ήταν ένας άνθρωπος του μέλλοντος, ο Χέλμουντ Κόλ. Για το γερμανικό λαό έφερε την εποχή της ενότητας. Και έχουμε μια νέα Γερμανία, όπου έχει μεγαλώσει ήδη μια νέα γενιά ανθρώπων σε αυτήν. Και το είπαν ήδη οι προλαλήσαντες. Τότε δεν ήταν όλοι έτοιμοι να το δεχτούν αυτό, αλλά ο Χέλμουτ Κόλ ήξερε πολύ καλά τι εστί πόλεμος. Το είχε δει ως έφηβος και χρειάστηκε πολύ καιρός για να καταφέρει η Ευρώπη να μην έχει χαρακόμματα και τύχη και εχθρικές ιδεολογίες που να την χωρίζουν. Ο Χέλμουτ Κόλ είχε αντιληφθεί πάρα πολύ καλά ότι Μόνο με αυτόν τον τρόπο, εάν ενωνόταν ολόκληρη η Ευρώπη, θα μπορούσε να ξαναενώσει την πατρίδα του. Σε αυτήν του την πορεία η Ρωσία, η χώρα μου, στάθηκε στο πλευρό του. Ο λαός μας αντιλαμβανόταν πάρα πολύ καλά τον κίνδυνο της σύγκρουσης και την αξία της ειρήνης. Αυτό επέτρεψε στους χθεσινούς εχθρούς να έχουν μία σχέση αμοιβαίου σεβασμού και ισότητας. Ο Χέλμουτ Κόλ προσωπικά έκανε πάρα πολλά ώστε οι σχέσεις μας να είναι οι καλύτερες που ήταν ποτέ στην ιστορία. Και αυτό η Ρωσία το εκτιμά ιδιαίτερος. Χέλμουτ Κόλ πέτυχε τον κύριο στόχο της ζωής του. Και πάντα παρέμενε ένας εθνικός ηγέτης, ο οποίος όμως σκεφτόταν και δρούσε σε ένα ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πλαίσιο. Δεν στόχευε μόνο στην Ενωμένη Γερμανία, αλλά στην Ενωμένη Ευρώπη και έβλεπε την Ρωσία ως μέρος αυτής. Στόχευε ακριβώς να δει μια Ήπειρο χωρίς αγκαθωτά σειρματοπλέγματα, χωρίς έχθρα. Μια Ευρωπαϊκή Ήπειρο ειρήνης και ασφάλειας για όλους. Όταν ένας άνθρωπος ξεπερνά τα κράτη και τα σύνορα και έχει τέτοιες ιδέες όπως η συνεργασία και η εμπιστοσύνη επιτυγχάνει τον στόχο του. Βεβαίως δεν μπορούμε να πούμε ότι τώρα η πορεία αυτή έχει τελειώσει, ότι έχουμε ένα ιδεώδες αποτέλεσμα. Πρέπει να παλεύουμε κάθε μέρα. Έπεσε το τείχος του Βερολίνου, και τώρα έχει κοπεί σε κομμάτια και το μοιράζουν σαν σουβενίρ. Αλλά πρέπει να παρατεχτούμε ότι σήμερα λόγω των αντιφάσεών μας απέχουμε πολύ από το να εφαρμόσουμε το όνειρο του κοινού σπιτιού μας, αλλά πρέπει να αντιληφθούμε ότι ενωμένοι, ασφαλείς και με ευημερία είναι η Ευρώπη την οποία θέλουμε. Ο Χέλμουτ Κόλ απέδειξε ότι ο στόχος αυτός μιας ενωμένης και ασφαλούς Ευρώπης είναι κάτι το οποίο μπορούμε να επιτύχουμε. Και αυτή είναι η ευθύνη που βαραίνει σήμερα τους ώμους όλων των Ευρωπαίων ηγετών. Κυρίες και κύριοι, η ζωή του καγκελαρίου της γερμανικής ενοποίησης θα παραμείνει στην μνήμη των ανθρώπων όλου του κόσμου. Στην Ρωσία θα τον θυμόμαστε ως έναν φίλο, έναν σοφό πολιτικό και έναν έξυπνο άνθρωπο. Έναν ανοιχτό και ειλικρινή άνθρωπο. Εξ ονόματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας θα ήθελα να εκφράσω τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια. Στους ε, συγγενείς του μεγάλου αυτού γιου της Γερμανίας, του Χέλμουτ Κόλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ τον κύριο Εμμανουέλ Μακρόν, πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, να εκφωνήσει την ομιλία του. Κυρία μου, μέλη της οικογένειας Κόλ. Κυρίες και κύριοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων, κυρίες και κύριοι υπουργοί, κυρίες και κύριοι πρέσβεις, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που διαλέξατε το Στρασβούργο ένα από τα μέρη, ένα από τους τόπους ορόσημα της Ευρώπης όπου τόσο πολύ αγάπησε ο κύριος Κόλ και έκανε τόσα για να ξαναβρισκόμαστε σήμερα εδώ. Επιτρέψτε μου να εκφράσω εδώ και μια σκέψη φορό για τη Σιμών Βέιλ. την γυναίκα αυτή που χάσαμε χθε, την πρώτη γυναίκα βουλευτή και έπειτα πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία ήξερε το τίμημα της Ευρώπης διότι είχε ζήσει την ε, ανίποτη και ανεξίτηλη εμπειρία του θανάτου. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ συγκεντρωμένοι για να τιμήσουμε τη μνήμη του Χέλμουντ Κόλ. Και περισσότερο από τη μνήμη του, το αποτύπωμα που έχει αφήσει στην ιστορία. Πολλοί από εσά με συγκίνηση αναφέρατε στιγμές που μοιραστήκατε μαζί του. Όμως για τη δική μου τη γενιά, ο Χέλμουτ Κόλ είναι ένα μέρος της ευρωπαϊκής ιστορίας. Είναι μια εμπειρία ζωής, ένα βίωμα που το ζούμε ακόμα. Μιλάμε για ιστορικές χειρονομίες, για πράξεις τόλμης ε, που έχουν γράψει ιστορία και χωρίς τις οποίες η δική μας γενιά δεν θα είχε κάνει τις, τις σωστές επιλογές. Εκατοντάδες σελίδες έχουν ε, γραφτεί για την προσφορά του Χέλμουτ Κόλ, για τη δράση του, την επανένωση της Γερμανίας και την οικοδόμηση της Ευρώπης. Τα έχετε αναφέρει διαμακρών όλοι. Είναι αυτός ο άνθρωπος που επανειλημμένος έλαβε τολμηρές αποφάσεις, πολλές φορές κατά την κοινή γνώμη της χώρας του. Πολλές φορές ε, ε, όταν δεν ήταν κάτι επιθυμητό ή που αναμενόταν αυτό που αποφάσιζε ως πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας θα ήθελε κληρονομιά του να μην ε, παραμείνει ένας πολιτικός απολογισμός το μάθημα που μας δίνει ο Χέλμουτ Κόλ ξεπερνάει τα όρια του πολιτικού απολογισμού που μένει στις σελίδες των απομνημονευμάτων. Ήταν ένας συνομιλητής της Γαλλίας προνομιακός ένας ε, άνθρωπος που έχτιζε άοκνα, αλλά πάνω από όλα ήταν φίλος της Γαλλίας. Η σχέση του με τη Γαλλία τροφοδοτεί το από την προσωπική, οικογενειακή και ιστορική του μνήμη ζυμώθηκε μέσα από την περιέργεια που ένιωθε αυτός ο άνθρωπο που γεννήθηκε στη Ρινανία και έστρεφε το βλέμμα προς του γειτονέ του πέρα από το ποτάμι που ε, μας κάνει γείτονες ε, αλλά και μας χώριζε. Προτιμούσε πάντοτε τις γέφυρες από τα τείχη και τα σύνορα. Αυτή η σχέση σημαδευόταν από τον ε, ανίποτο σεβασμό που τον έφερνε αντιμέτωπο με τους φανατισμούς και την αγριότητα, την σκληρότητα της βίας. Όταν στις αρχές της δεκαετίας του 80 οι Γάλλοι επέλεξαν πολιτικούς ηθήνοντες των οποίων οι οικονομικές επιλογές αναστάτωναν κάποιους από τους εταίρους μας, ο Χέλμουτ Κόλ μας έτεινε τη χείρα της συνεργασίας, ξεπερνώντας τις επιφυλάξεις κάποιων από τους πολιτικούς του φίλους. Ε, έπειτα όταν ε, μας δίχασαν σε σχέση με το θέμα της Ευρώπης κυρίως οι εθνικές μας απόψεις, οι εσωτερικέ μα απόψει, επιβεβαίωσε την εμπιστοσύνη του σε εμά. και όταν ανησύχησε του άλλου η ε, επανένωση τη Γερμανία, ε, κατέβαλε κάθε προσπάθεια για να μην αποδυναμωθεί η Ευρώπη αλλά να ενισχυθεί μέσα από την επανένωση της Γερμανίας. Η Γαλλία φάνηκε αντάξια αυτής της φιλίας που ε, ήταν αμύωτη στο χρόνο. Μετά τον Σάρλ Ντεγκόλ, τον Κορτάν τον Βαλέντι Ζεσκάρντεσταν και τον Χέλμουντ Σπίτ που είχαν τα θεμέλια της Ευρώπης, ο Φρανσουά Μιτερό πήρε την ε, σκητάλη από αυτούς ε, μαζί με τον Χελμουτ Κόλ. Και ο ένας και ο άλλος μπόρεσαν να ξεπεράσουν τις τραγικές εμπειρίες της γενιάς τους. Και ο ένας και ο άλλος υπέφεραν επειδή οι λαοί τους ήρθαν αντιμέτωποι και συγκρούστηκαν. Ε, λαοί που θα μπορούσαν να είναι φίλοι. Έτσι, ο Χέλμουντ Κόλ και ο Φρανσουά Μιτερά μετά και ο Ζακ Σιράκ έδειξαν με έγκλη ότι η Ευρώπη είναι μεγάλη και ισχυρή. Μόνο αν είναι μεγάλη και ισχυρή η καλή ε, προαίρεση και η φιλία στην οποία βασίζεται η σχέση τους η σχέση των κρατών. Στις 4 Ιανουαρίου 1990 ο Χέλμουτ Κόλ επισκέφθηκε τον Φρασουά Μιτερόν στην κατοικία του στο Λατσέ. Μετά από πολλές συζητή... εβδομάδες συζητήσεων για την επανένωση της Γερμανίας, αυτή η επίσκεψη επέτρεψε σε αυτούς τους δύο άντρες να συζητήσουν όλα τα θέματα ε, που τους απασχολούσαν ε, στα ε, ε, στην άμμο αυτής της περιοχής της Γαλλίας, της Λόντ, μέσα στα Πεύκα. Αυτή η συντροφιά δύο περεπατητών ήταν που τους ε, ε, ένωσε ακόμη περισσότερο. Και έτσι γράφεται κάποιες φορές το πεπρωμένο του κόσμου, με την μοίρα δυο ανθρώπων. Ο Χέλμουτ Κόλ και ο Φρανσουά Μιτερό έδειξαν ότι η αδερφοσύνη μπορεί να γίνει μόνο ε, να αποκτήσει νόημα όταν ενώνει πραγματικά τους ανθρώπους. Πρέπει αυτό να φανεί και στα θεσμικά όργανα και στις συμφωνίες. Και πήραν οι ίδιοι το ρίσκο, ανέλαβαν το ρίσκο να επιβεβαιώσουν αυτή τη φιλία σε επίπεδο θεσμών και συμφωνιών. Αυτή η ε, δράση λοιπόν ε, του Helmut Kohl άφησε το αποτύπωμα χωρίς προηγούμενο και μας φέρνει εδώ σήμερα. Οι ευρωπαϊκές συνθήκες πολλές φορές και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί ε, αντιμετωπίζονται ως κενά δημιουργήματα από πολλούς και επικρίνονται. Θέλω να πω μπροστά στον Χέλμουτ Κόλ ότι επειδή δεν ε, νιώθετε πια την φιλία που σας ενώνει, επειδή εσείς αφήνατε να πεθάνει αυτή η φλόγα που έχτισε τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τις συνθήκες. Επειδή ξεχάσατε τη μοίρα στην οποία ε, θεμελιώθηκαν, γι' αυτό είναι κενά νοήματος. Επειδή ε, ε εσείς ε, αποφασίσατε η Ευρώπη να είναι τεχνοκρατική, είναι έτσι. Αλλά ποιο ήταν το μήνυμα της ζωής, το αποτύπωμα και το ίχνος του προμένου του Χέλμουτ Κόλ ήταν να μας δείξει ότι η Ευρώπη μας, αυτή που μας ενώνει σήμερα, είναι καρπός της προσπάθειας και της ιστορίας πολλών γενεών πολλών πεπρωμένων, πολλών ανθρώπων που αποφάσισαν να ξεπεράσουν τα όρια του πεπρωμένου τους και της μοίρας τους, που, που είχαν την τόλμη να υψώσουν το ανάστημά τους και να ξεπεράσουν το μίσος και το φόβο. Ποιο οικοδόμημα δεν χάνει το νόημά του και την ομορφιά του εάν δεν κατοικείται πλέον από κανέναν. Αυτό είναι το μάθημα που μας αφήνει ο Χέλμουτ Κόλ ε, στη Γαλλία και σε όλους τους Ευρωπαίους είναι ότι ο πραγματισμός, ο ρεαλισμός, η πολιτική επιδεξιότητα είναι πολύ χρήσιμα στοιχεία, όμως δεν χτίζουν τίποτα από μόνα τους. Είναι τα ιδεώδη και τα ιδανικά που τα φωτίζει η φιλία και ο πλούτος μια ζωής που δίνουν σάρκα και οστά σε ένα εγχείρημα, που το επιτρέπουν να έχει διάρκεια ζωής. Με αυτά τα στοιχεία η Άγγελα Μέρκελ και εγώ θέλουμε να δώσουμε ένα νόημα λογική και ε, μια πορεία στην Ευρώπη. Η ιστορία κάποια μέρα θα κρίνει και εμάς και θα σταθμίσει με αυστηρότητα τις παραχωρήσεις που ενδεχομένως τα έχουμε κάνει προς όφελος κοντόφθαλμων υπολογισμών ή εθνικιστικών εγωισμών ή στην ευκολία της στιγμής. Αυτό όμω που θα μετρήσει υπέρ μα θα είναι η ειλικρίνεια με την οποία αφοσιωθήκαμε στην ειρήνη και την ομόνια μεταξύ των λαών. Θα είναι η αφοσίωσή μα ε, στο ευρωπαϊκό αυτό εγχείρημα που είναι προπόθεση για την ομόνια και την ειρήνη μεταξύ των λαών. Για τη βαθιά φιλία που ξεκινάει από την κοινή μα ιστορία, από του πολιτισμού μα που είναι τόσο στενά αλληλένδετοι και από τι κοινέ δοκιμασίε που έχουμε περάσει όλοι λέει. Και αν κάποιε φορέ ε, μα κυριεύει η αμφιβολία σε αυτό το τιτάνιο καθήκον, Λοιπόν, πρέπει απλώ να σκεφτούμε τη μεγάλη φυσιογνωμία του Χέλμουτ Κόλ και να το αποτίσουμε φορό με την ευγνωμοσύνη που του οφείλουμε. Να θυμηθούμε αυτή την έκφραση που ε, ανακεφαλαιώνει όλη του τη ζωή. Σήμερα δεν έχουμε κανένα λόγο να παρατηθούμε από τις προσπάθειές μας. Έχουμε πολύ περισσότερους λόγους να είμαστε ρεαλιστικά αισιόδοξοι. Για πολύ καιρό ακόμα θα αντλούμε μαθήματα από την υποδειγματική του ζωή. Ό,τι χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την κοινή μας πορεία. Κυρίως την τόλμη και την ελπίδα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας. Και τώρα θα ήθελα να παρακαλέσω την κυρία Δόκτωρα Αγγέλα Μέρκελ, καγκελάριο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας Γερμανίας, να λάβει το λόγο. Αξιότιμοι Πρόεδροι και Πρωθυπουργοί, εξοχότατοι αξιότιμοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Αγαπητή κυρία Κόλ Ρίχτερ, αγαπητή οικογένεια Κόλ. Σήμερα αποχαιρετούμε τον Χέλμουτ Κόλ, τον καγκελάριο της Γερμανικής Επανένωσης, κάτοχο βραβείο Καλομάγνου και επίτιμο πολίτη της Ευρώπης. Εκείνος που σπούδασε ιστορία όταν ήταν νέος, έχει βρει ο ίδιος τη θέση του στα ιστορικά εγχειρίδια. Ο Χέλμουτ Κόλ ενσαρκώνει μια ολόκληρη εποχή με την εσωτερική και εξωτερική πολιτική άνοιξε δρόμους που ισχύουν ακόμα. Η θητεία του συνδέεται με πολλά χρόνια οικονομικής ευμάρειας, αλλά παρόλα αυτά δεν έχασε ποτέ την εικόνα τη συνολική, πέρα από τη Γερμανία και πέρα από την εκάστοτε ημέρα. Συνδιαμόρφωσε ρηξικέλευτες αλλαγές και συνδημιούργησε αποφασιστικά την Ευρώπη και την Γερμανία στην οποία σήμερα ζούμε. Πολλά από αυτά που σήμερα για μας είναι αυτονόητα ανάγονται σε εκείνον. Η Ενωμένη Δυτική και Ανατολική Γερμανία, η ενιαία αγορά, η κατάργηση των συνόρων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γεγονός ότι τα περισσότερα κράτη της Ένωσης έχουν το ίδιο νόμισμα το γεγονό ότι υπάρχει καν η Ευρωπαϊκή Ένωση υπό τη σημερινή τη μορφή, όλα αυτά είναι και παραμένουν συνδεδεμένα άρρηκτα με το όνομα του Helmut Κόλ. Έχει σφραγίσει μια ολόκληρη γενιά. Πολλοί συγκρούστηκαν μαζί του και υπήρξαν και προστριβές. Πολλοί μπορούμε να σας διηγηθούμε περιστατικά και εγώ προσωπικά, αλλά όλα αυτά είναι σε δεύτερη μοίρα μπροστά στο τεράστιο έργο του. Και αυτό και οι πολιτικοί του αντίπαλοι των τιμούν και το σέβονται. Πώς εξηγείται. Αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση προσωπικά στο Helmut Kohl ήταν η εξαιρετική αίσθηση που είχε για το πολιτικά εφικτό αλλά και η ακράδαντη πεποίθησή του και αυτό δεν είναι αντίφαση ε, που πριτάνευε κάθε φορά στις αποφάσεις του μπορούσε κανείς να υπολογίζει στο Helmut Kohl. Από την αρχή επέλεγε στελέχη να το πλαισιώνουν, ε, πράγμα που εξέπλητε και άφηνε και μεγάλη ελευθερία στα στελέχη που το πλαισίωναν. Είχα την ευκαιρία να το διαπιστώσω και εγώ προσωπικά. Και βέβαια δεν ήταν πάντα εύκολο ε, να ε, περάσει κανείς τα επιχειρήματά του δεν ήταν εύκολο, αλλά πάντα ήταν στο πλευρό και συμβούλευε και άκουγε τους συνεργάτες του σε πολύ συγκεκριμένες φάσεις της ζωής. Όπως το 1992 επί σειράμενων, ε, να μπορέσω να ε, συνδυάσω ε, τη θέση μου ως υπουργό με ένα κάταγμα που με ταλαιπώρησε πάρα πολύ καιρό, κάταγμα στο πόδι. Είχε και ανθρώπινες σχέσεις και στενές φιλίες και στη Γερμανία και στην Ευρώπη και παγκοσμίως κατάφερε να σφυριλατήσει αξιόπιστες σχέσεις, ε, να ε, κάνει φιλίες και να συνεργάζεται. Ήταν ένας παγκόσμιος πολιτικός στραμμένος προς τους ανθρώπους. Όταν ανέλαβε ε, καγκελάριο το 1982. Η πρώτη επίσκεψή του ήταν στο Παρίσι. Ένα σύμβουλο του Προέδρου μητέρα, ε, στη συνέχεια είπε ότι αρχικά οι Γάλλοι ήταν πολύ επιφυλακτική, αλλά μετά και παραπέμπω, ε, αμέσως ήμασταν ε, πάρα πολύ ενθουσιώδεις και φλογεροί. Αυτό ενσάρκωνε και τη γαλλογερμανική φιλία. Βαθιά στη μνήμη των εθνών μας, έχει καταγραφεί η εικόνα των δύο ηγετών ε, στο Βεχντά, μπροστά στα χαρακόμματα, χέρι-χέρι. Αυτό ως χειρονομία συμφιλίωσης και ενότητας σφράγισε ένα νέο κεφάλαιο κοινή ιστορίας. Ήξερε να χτίζει γέφυρες. Μέχρι το Παρίσι, μέχρι τη Βαρσοβία, μέχρι την Ουάσιγκτον και τη Μόσχα έφταναν. άοκνα εργαζόταν με τους ε, συνεργάτες και με τους εταίρους. Ως παιδί και νέος έζησε ο ίδιος τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ανίποτο, ε, φρικτό και τα δεινά που είχε φέρει η Γερμανία και ο εθνικοσοσιαλισμός στην Ευρώπη και στον κόσμο. Αλλά και τις αγωνίες και το φόβο στους νυχτερινούς βομβαρδισμούς. Ακριβώς αυτές οι εμπειρίες και τα βιώματα τον οδήγησαν να συμμετέχει νέος και να δεσμευτεί στο νέο κόμμα τότε της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης. Γι' αυτό είχε και το αξίωμα για την εξωτερική πολιτική που δεν χωρούσε αμφισβητήσεις και αμφιβολίες. Θα πρέπει να αγωνιστούμε για μια ισχυρή Ευρώπη που δεν θα υπάρχουν ποτέ πια πόλεμοι. Αυτός ο στοχασμός και αυτή η σκέψη που ήταν ενταγμένη στο ε, ιστορικό γίγνεσθε τον καθόρισε. Ταυτόχρονα όμως ήταν προσιλωμένος ε, την πατρίδα του, όλη του τη ζωή, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο Παλατινάτο, με βαθιές ρίζες εδώ στην περιφέρεια, στην κεντρική Ευρώπη. Αλλά καταλάβαινε πολύ ε, την αίσθηση και τη σκέψη των γειτόνων. Αυτό το καταλάβαιναν, το ένιωθαν οι συνομιλητές, ήξεραν ότι μπορούν να υπολογίζουν σε εκείνον. Ό,τι έλεγε το ε, υποστήριζε και σε ό,τι δεσμευόταν. Ανεπιφύλακτα όταν ανέλαβε καγκελάριο, η Γερμανία και η Ευρώπη ήταν διχασμένες. Με ένοπλη ε, αντιπαράθεση και σύραξη να παραμένει ένα φάντασμα και ένα σενάριο τρόμου. Στο τέλος της θητείας του, η ε, ε, Γερμανία ήταν ενωμένη και για πρώτη φορά στην ιστορία συμφιλειωμένη και εν ειρήνη, φιλία και συνεργασία με όλους τους γείτονες εργάστηκε για τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ προς ε, την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και προετοίμασε το έδαφος. Είχε αποφασίσει και το νέο νόμισμα. Όταν ανέλαβε το 1982 ο Χέλμουτ Κόλεγο ζούσα στην Ανατολική Γερμανία. Και άκουσα στην τηλεόραση και είδα το 1987 την ομιλία του με το Χόνεκερ στη Βόνη. Όταν είπε ο Χόνεκερ, οι άνθρωποι από τη Γερμανία, μάλλον είπε στο Χόνεκερ, ότι ζουν οι άνθρωποι ενωμένοι, αλλά στη Γερμανία διχασμένοι. Θα πρέπει ε, να ρίξουμε αυτό το τείχος. Οι άνθρωποι θέλουν να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα, διότι ε, θα πρέπει να ζουν μαζί. Αυτά τα λόγια είπε στο Χόνεκερ και αυτό μας έδωσε δύναμη στην Ανατολική Γερμανία. Στη Πολωνία και σε άλλες χώρες τα κινήματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο νέος άνεμος που έπνεε από τη Μόσχα μας έδιναν και μας θάρρος στην Ανατολική Γερμανία. Εκατοντάδες χιλιάδες τόλμησαν να βγουν στο δρόμο και διαδήλωσαν για την ελευθερία και κατάφεραν να ρίξουν το τείχος. Και ο Χέμουτ Κόλ ήταν εκείνος ο οποίος ήθελε την ενότητα και την επανένωση όταν κάποιοι αμφέβαλαν ή ε, διαφωνούσαν. Ανέκαθεν σκεφτόταν τα συμφέροντα και των γειτόνων και των εταίρων μας. Ήταν ακράδαντα πεπισμένος Ευρωπαίος. Και πάντα ανησυχούσε και σκεφτότανε τι θα σήμαινε μια ε, Ενωμένη Γερμανία και κατάφερε να διασκεδάσει τους φόβους και τις αμφιβολίες των γειτόνων και φίλων μας. Αυτό θα παραμείνει ως μοναδική ιστορική κατάκτηση. Μαζί με τους εταίρους και συνεργάτες κατάφερε να εγγράψει την ενοποίηση της Γερμανίας στην Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Αυτό ήταν έργο ειρήνης, ήταν έργο ενότητας. Ο Άντεναορ, ο Ζαμονέ, ο Ρομπέρ Σουμάν και άλλοι συναντούν εδώ τον Χέλμουτ Κόλ η Ευρώπη είναι έργο γενεών. Κάθε γενεά έχει τις δικές της προκλήσεις να αντιμετωπίσει. Κάθε γενεά θα πρέπει να βρει τις δικές της απαντήσεις για το πώς θα θωρακίσει την Ευρώπη για το μέλλον. Και κάθε φορά αυτό που διακυβεύεται είναι εκείνο που ήξερε ο Χέλμουτ Κόλ. Να γνωρίζεις την ιστορία, να βλέπεις μακριά και σε μεγάλο χρονικό ορίζοντα, αλλά να είσαι κοντά στους ανθρώπους να έχεις αίσθηση του εφικτού και τι μπορεί να επιβάλλει στους άλλους. Υπάρχει ένα μνημείο στο κέντρο του Βερολίνου για τους Εβραίους που έχασαν τη ζωή τους. Και εκεί παραθέτουν κάτι που έχει ε, κάτι το χαρακτηριστικό για το έργο του Χέλμουντ Κόλ. Δεν είναι η επόμενη γενιά, αλλά η δική μας εκείνη που θα πρέπει να χτίσει. Εμείς, εδώ, τώρα, σήμερα και όχι κάποιος, κάποια στιγμή. Έτσι και αποφασίστηκε στη Γερμανική Βουλή με πλειοψηφία δύο τρίτων. Κυρίε και κύριοι, στη συνέχεια θα συνοδεύσουμε προς τη Γερμανία ξανά, το Χέλμοντ Κόλ. Θα περάσει από την πόλη που γεννήθηκε, το Λούτβιξ Χάφον. Το σπίτι του ήταν εδώ. Πολλά χρόνια με την πρώτη του σύζυγο Χάνε Λόρε, που ήταν πάντα στο πλευρό του, σε καλού και χαλεπού καιρού. Και σε εκείνη αποδίδουμε με φοροτιμή ευγνωμονώντε. Και κυρία Κόλ Ρίχτερ, εσεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια με αυταπάρνηση και με αγάπη συνοδεύσατε το σύζυγό σας μέχρι τελευταία στιγμή. Τα συλληπιτήριά μου και τα συλληπιτήριά μου και προς όλους άλλους στην οικογένειά του που τον πενθούν σήμερα. Στη Σπάιερ θα κλείσει η σημερινή ημέρα και πάλι θα κλείσει ο κύκλος από τη Γαλλία προς τη Γερμανία, στην Πατρίδα, στο Παλατινάτο. Από επίτιμος πολίτης Ευρώπης, καγκελάριος της Γερμανικής Ενοποίησης. Έτσι θα τον θυμόμαστε όλοι. Χωρίς τον Χέλμουτ Κόλ, η ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων μέχρι το, που ζούσαν μέχρι το 1990 πίσω από το τείχος θα ήταν τελείως διαφορετική. Φυσικά και η δική μου. Αγαπητέ καγκελάρι Χέλμουτ Κόλ, το γεγονός ότι βρίσκομαι εγώ σήμερα εδώ έχει να κάνει και με εσά. Ήταν σημαντική η συνεισφορά Σα Σα ευχαριστώ για τι ευκαιρίε που μου δώσατε. Σα ευχαριστώ για τι ευκαιρίε που δώσατε και ανοίξατε σε πολλού άλλου. Σα ευχαριστώ για τι ευκαιρίε που έχουμε εμεί ω Γερμανοί και ω Ευρωπαίοι, χάρη σε εσά. Έχετε επιτύχει άπειρα πράγματα. Α αναπευθείτε εν ειρήνη. Τώρα είναι η σειρά μα να διατηρήσουμε και να διαφυλάξουμε την κληρονομιά σας γονατίζω μπροστά σας και στη μνήμη σας ευγνωμονούσα και με ταπεινότητα. Ευχαριστώ πολύ, Καγκελάρη.